Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την κατεπίγουσα βοήθεια των προσφύγων και μεταναστών που έχουν προβλήματα αγωσκοκαιρία στα, στα τόπεδα της Ευρώπης. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Μπόργκα ε, που θα μιλήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου. Grazie. Onorevoli membri, Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη. Η ανησυχία σας για την κατάσταση και τη μοίρα των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που αντιμετωπίζουν σοβαρές καιρικές συνθήκες στους ευρωπαϊκούς καταβλισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν οι ελληνικές αρχές, πάνω από 15.000 μετανάστες είναι παρόντες στα ελληνικά νησιά. Τα hot spots, τα σημεία υποδοχή, ε, πάσχουν από πληθυσμό και οι συνθήκε διαβίωση είναι δυσχερέστατε λόγω των συνθήκων των χειμερινών. Έτσι δε περαιτέρω, η πατερμοστία του ΙΕ για πρόσφυγε λέει ότι 7.000 πρόσφυγε έχουν απομονωθεί στη Σερβία. Κάποιοι από αυτού παραμένουν σε στιμωγμένε συνθήκε ε, στο κέντρο του Βελιγραδίου. Ε, Βεβαίω δεν μπορούμε να αλλάξουμε τι καιρικέ συνθήκε αλλά έχουμε στη διάθεσή μας πόρους και εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να διορθώσουν τις άμεσες αρνητικές συνέπειες ε, των σοβαρών καιρικών συνθήκων. Ο Επίτροπος θα σε ενημερώσει όσον αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη χρήση της κατεπίγουσας χρηματοδότησης για να μειωθούν τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα καθώς και άλλες μορφές υποστήριξης που ήδη παρέχονται για τις πιο πλέον πληγήσεις χώρες και κάτι που προβλέπεται. Θα ήθελα λοιπόν, αν επιτρέπετε, να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου στα Μαλτέζικα. Έχουμε επίγνωση του ότι οι ελληνικές αρχές έχουν στείλει ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού στη Λέσβο για να βοηθήσει τους μετανάστες εκείνους που αντιμετωπίζουν αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η Προεδρία μας παρακολουθεί εκ του σύνεγγης την όλη κατάσταση, ταυτόχρονα γνωρίζει και είναι σε επαφή με όλες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες του τομέα. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, ούτω ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες καθώς και να μειώσουμε και ίσως τα προβλήματα και να τα λύσουμε ίσως. Οι υποχρεώσεις που ανελήφθησαν όσον αφορά την παροχή μέτρων ε, κέντρων υποδοχής που θα προσαρμόσουν το χειμώνα θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν ταχύτερο δυνατόν. Καμία χώρα δεν ε, μπορεί να ελέγξει την κατάσταση από μόνη της. Αλλά η δουλειά μας δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο από τις χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή του προβλήματος και άλλες χώρες πρέπει να παράσουν υποστήριξη. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε την κατάσταση κατά την οποία ε, επιδεινώνονται, το, τα προβλήματα μέσω ενιαίας προσέγγισης και αλληλεγγύης. Και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα και θα πρέπει και να έχουμε κάποια σχέδια μακροπρόθεσμα. Μία από τις προτεραιότητες για το εξάμεινό μας είναι να ενθαρρύνουμε την εφαρμογή σειράς μέτρων που ήδη έχουμε συμφωνήσει και να εξασφαλίσουμε το ότι τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται θα είναι στο θεματολόγιο που θα συζητείτε. Αυτό αναφέρθηκε το πρωί εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας από τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Τζόσεφ Μουσκάτ. Όπως γνωρίζετε, προεδρεύουμε του Συμβουλίου σε αυτή τη φάση και περιμένουν οι πολίτες να κάνουμε κάτι, κάποια δράση από μας η μεταγκατάσταση μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να μειωθούν οι συνέπειες της κρίσης. Όμως, ακόμα και αν υπήρξε πρόοδος που έχει καταγραφεί, αυτή η πρόοδος είναι αργή. Μέχρι τις 11 πρώτου Ιανουαρίου, περίπου 8.000 άνθρωποι έχουν μεταγκατασταθεί στην Ελλάδα. Αν επιταχύνουμε την όλη διαδικασία, θα βοηθήσουμε και την Ελλάδα και αυτό θα έχει και τεράστιο αντίκτυπο για τη ζωή των προσφύγων. Αιτήσει για μετεγκατάσταση θα πρέπει να αυξηθούν και μάλιστα κατεπηγόντως και τα κράτη-μέλη θα πρέπει γρήγορα να απαντήσουν θετικά για τη μετεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων μέχρι τον αρμοδι... μέσω των αρμοδίων φορέων της Frontex και της EASO, βοηθώντας έτσι τα κράτη-μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν άμεσα αυτή την κρίση. Αυτό είναι κάτι που θα απαιτεί τότε ώστε να επιταχυνθεί η εφαρμογή της διαδικασίας κατάσταση των προσφύγων. Μακροπρόθεσμα η σταθερότητα όσον αφορά τον, τον ανατολικό διάδρομο είναι κάτι που απαιτείται. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια στη Μεσόγειο, χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ενώσεω, χρειαζόμαστε περισσότερε δεσμεύσει για τη βελτίωση των διαδικασιών, για τι αιτήσει ασύλου, καθώ και για τι επιστροφέ μεταναστών προς την Τουρκία. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία ε, όσον αφορά τις χώρες της, ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό είναι κρίσιμο. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξετάσουμε τις νομοθετικές προτάσεις για μεταρρύθμιση για ένα κοινό σύστημα, ευρωπαϊκό κοινό σύστημα ασύλου, ούτω ώστε να συνεχίσουμε την εργασία προηγούμενων προεδριών της ε, Ολλανδικής ε, Προεδρίας και της απερχόμενης Σλοβακικής, ούτως ώστε να έχουμε ε, μία συνέχεια και η συνεργασία ε, να υποδιαιρείται με καλύτερο, πιο δίκαιο τρόπο. Στο τέλος θέλουμε κυρίες και κύριοι να έχουμε μια βιώσιμη πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση και το, και το άσυλο και αυτό χρειάζεται και περισσότερους ελέγχους στα σύνορά μας θα πρέπει να επιλύσουμε και κατεπήγοντα προβλήματα όπως αυτά που συζητούμε σήμερα ούτως ώστε να διασώσουμε ζωές και να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα που θα εφαρμόζουμε θα είναι δίκαιο. Εκτιμήσουμε πολύ τη βοήθειά σας. Είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο τον κύριο Στυλιανίδη, τον Επίτροπο. Αγαπητή κυρία... αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί υπουργοί. Σας ευχαριστώ για αυτή την επίκαιρη συζήτηση. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τις σκληρότερες χειμερινές συνθήκες που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι το, τη Βόρεια Ευρώπη. Σε ορισμένα μέρη μάλιστα της Ευρώπης αυτό δεν ήταν ε, αναμενόμενο, αλλά Όλοι μας είδαμε τις εικόνες στον τύπο για πολλούς, που αφορούσαν πολλούς καταβλισμούς προσφύγων. Θα είμαι σαφής, κανένας δεν είναι περήφανος για αυτή την κατάσταση. Η ηθική μας υποχρέωση είναι προσφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο αξιοπρέπεια σήμερα. Όχι την επόμενη εβδομάδα, όχι αύριο. Γι' αυτό βοηθάμε τις αρχές ε, στην ε, αντίδρασή τους, στην ανταπόκρισή τους σε όλες τις επίγουσες ε, δράσεις τις οποίες πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα ώστε να επιταχυνθεί η προσαρμογή στο χειμώνα στους καταβλισμούς. Ο αγαπητός συνάδελφος Επίτροπος Αβραμόπουλος και εγώ είμαστε σε τακτική επαφή με τις ελληνικές αρχές στα ελληνικά νησιά όπου η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή διερευνούμε όλες τις δυνατές λύσεις ώστε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ήταν στη Λέσβο νωρίτερα σήμερα ώστε να μπορέσει διεισόμαστε να αξιολογήσει την κατάσταση επιτόπου και βεβαίως να συζητήσει και να βρει άμεσα λύσεις. Καλωσορίζουμε την γρήγορη ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστεί η δύσκολη κατάσταση στα νησιά. Πρώτον, για μετακίνηση των πιο ευάλωτων σε χώρους υποδοχής ανθεκτικούς σε χειμερινές συνθήκες. Δεύτερον, να διεκπαιρεώσει γρήγορα τις διαδικασίες ασύλου για τους ανθρώπους, ε, ιδιαίτερα τους ευάλωτους που μπορούν να επιστραφούν στην Τουρκία και έπειτα να χρησιμοποιήσει πλοία του στρατιωτικού ναυτικού ώστε να ε, στεγαστούν ε, όσοι είχαν ε, ανάγκη, ιδιαίτερα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες. Συζητάμε δε την δημιουργία κατάλληλων ε, καταφυγίων, ε, καταλημάτων στα νησιά, αλλά και τη δυνατότητα βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών. Όπως ο αγαπητός συνάδελφος ε, Αβραμόπουλος ε, μου ανέφερε και είπε σήμερα και στη Λέσβο ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν μόνο σε συνεργασία και με τη στήριξη των τοπικών αρχών. Και βεβαίως με την στήριξη των τοπικών ε, πληθυσμών στα νησιά που έχουν ε, επιδείξει τεράστια γενοδορία απέναντι στις εκατοντάδες και χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν ε, φυγθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε έτοιμοι ώστε να παράσχουμε χρηματοδότηση για να δημιουργηθούν οι επιπλέον ε, τα επιπλέον καταλήματα και αυτό το έχουμε ε, ανακοινώσει στις, αρχές, στις εθνικές και τοπικές αρχές. Ε, το ίδιο κάνουμε και στην υπηρετική Ελλάδα σε συνεργασία με το UNHCR και με άλλους εταίρους ανθρωπιστικής βοήθειας. Η διάφοροι εταίροι ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης, ε, οι διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ, ΜΚΟ, είναι επιτόπου, βοηθούν πάνω από 200.000 δε ε, αντικείμενα για την αντιμετώπιση του χειμώνα έχουν διανεμηθεί στους πρόσφυγες sleeping bag, υπνόσακι δηλαδή, ε, κουβέρτες, ζεστά ρούχα, Βεβαίω, αυτέ δεν είναι μακροπρόθεσμες λύσεις, αλλά αυτές οι έκτακτες καιρικέ συνθήκες απαιτούν και έκτακτες απαντήσεις. Παρακολουθούμε την κατάσταση στο νησιά, στο νησί ε, στενά και θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί ε, για να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές ε, για όσο καιρό αυτό χρειαστεί. Τώρα, για την υπηρετική χώρα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική είναι υποέλεγχο η αντιμετώπιση του χειμώνα. 31 ε, 31 ένας χώροι είναι εξοπλισμένοι για ε, χειμερινές συνθήκες και δίνεται και επίγουσα βοήθεια που είναι δική μου ευθύνη και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας γιατί έτσι φτιάξαμε αυτό το σύστημα και το διαχειρίζεται η DGI.com και οι δικές μου υπηρεσίες 200 εκατομμύρια δόθηκαν πέρυσι μόνο στον ανθρωπιστικό τομέα και το 25% του ποσού αυτού, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν σε εταίρους ανθρωπιστικής βοήθειας για να εξοπλίσουν τους χώρους ε, ε, για να αντιμετωπίσουν χειμερινές συνθήκες, ε, για να βελτιωθούν οι υγειονομικές συνθήκες, ε, να προσφερθεί θέρμανση και ούτω καθεξής. Είναι μακρύς ο κατάλογος και αυτό επιπλέον των κονδυλίων που ήδη είχαν διατεθεί από την αρχή του 2015 352 εκατομμύρια ευρώ ε, επίγουσες βοήθειας από τα κονδύλια εσωτερικών υποθέσεων δόθηκαν στην Ελλάδα. Αυτή η βοήθεια δόθηκε είτε άμεσα στις εθνικές αρχές είτε στις ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τους διεθνείς ε, οργανώσεις με στόχο την άμεση στήριξη της διαχείρισης ε, της μετανάστευσης στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης ε, της βελτίωσης των δυνατοτήτων υποδοχής καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση στου καταβλισμού τόσο στην υπηρετική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Αυτή η επίγουσα χρηματοδότηση συμπληρώνει τα 509 εκατομμύρια ευρώ που ήδη είχαν διατεθεί στην Ελλάδα υπό τα εθνικά προγράμματα για, το 2000, για την περίοδο 2014 μέχρι 2020 και εδώ να σας θυμίσω ότι στο, στο σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει πάνω από ένα δις ευρώ στην Ελλάδα υπό τα κονδύλια εσωτερικών υποθέσεων και το νέο μέσο ε, πήγουσας ε, υποστήριξης. Είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος αυτού, του, αυτών των κονδυλίων η Ελλάδα. Να στραφώ τώρα στην Σερβία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Κομισιόν χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσει τη χώρα αυτή να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση, όχι μόνο διότι αυτές οι δύο χώρες είναι υποψήφιες, αλλά ε, εδώ παρέχουμε σημαντική οικονομική και τεχνική στήριξη. Γνωρίζω τις τεράστιες δυσκολίες που οφείλονται στο ψύχος και τις ε, πολύ ε, ισχυρέ χιονοπτώσει στη Σερβία κυρίως και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο θα μεταβώ στη χώρα για να αξιολογήσουμε την κατάσταση επιτόπου και να συζητήσουμε με τις αρμόδιες αρχές, να συναντήσουμε τους πρόσφυγες και να εκφράσουμε και ακόμα μια φορά την απτή αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επεκτείνοντα τι δυνατότητε υποδοχή και εξασφαλίζοντα ότι οι καταβλισμοί που υπάρχουν ε, θα είναι προτεραιότητα για μας. Ε, 43 εκατομμύρια έχουμε δώσει στο Σερβία από τον Οκτώβριο του 2015 μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και της πενταξιακής βοήθειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έτσι ε, καθίσταται ο μεγαλύτερος δωρητής. 19 εκατομμύρια ανθρωπιστικής βοήθειας χορηγήθηκαν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής για χειμερινό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων για την παροχή ζεστών γευμάτων ε, άρα άλλα 24 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν μέσω του προενταξιακού μέσου βοηθούν επίσης τη Σερβία να φιλοξενήσει και να στεγάσει αυτούς τους μετανάστες και πρόσφυγες και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις δυνατότητές της ελέγχου των συνόρων της. Αυτά είναι κομμάτι πάνω από 118 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται από την Ένωση στο πλαίσιο της οικονομικής και τεχνικής στήριξης στον τομέα αυτό από το 2007. Βεβαίως, περισσότερα πρέπει να γίνουν ώστε να ε, υπάρχουν ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες για τους μετανάστες μέσω της επέκτασης και μέσω της επέκτασης των συνθήκων υποδοχής. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και γι' αυτό και θα μεταβώ στη χώρα αυτή το Σαββατοκύριακο ώστε να συζητήσω με τις σερβικές αρχές για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση επιτόπου. Στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας η χώρα αυτή φιλοξενεί γύρω στους 200 πρόσφυγες από τότε που ξέσπασε η κρίση το 2015 η Κομισιόν έχει χορηγήσει 19 εκατομμύρια ευρώ ώστε να βοηθήσει συγκεκριμένα την χώρα αυτή να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση συμπεριλαμβανομένης ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι κομμάτι των 50 εκατομμυρίων ευρώ ε, οικονομικής και τεχνικής στήριξης προς τη χώρα από το 2007 στο πλαίσιο των συνόρων της μετανάστευσης και της ε, ε, διαχείριση του ασύλου. Θα εξετάσουμε επιπλέον μορφές βοήθειας ε, καθώς θα προκύπτουν περαιτέρω ανάγκες. Αυτή είναι η κατάσταση στις τρεις ε, χώρες, Ελλάδα, Σερβία και Φύρομ. Και βεβαίως θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν είμαστε περήφανοι για αυτή την πολύ αδυνηρή κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε αρκετά χρήματα αλλά ορισμένες αδυναμίες επιτόπου δεν επέτρεψαν τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η άνευ κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο κύριος Δίας για δύο λεπτά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας συγχαίρω που, γιατί λάβατε και πάλι την εμπιστοσύνη της Ολομέλειας. Η Ευρώπη περνά ένα κύμα ψύχους ε, ε, χειρότερο ε, που έχουμε δει εδώ και πολλά δεκαετία, πολλές δεκαετίες και αυτό επηρεάζει τον κόσμο που βρίσκεται στα σύνορα των Βαλκανίων και χτυπά περισσότερο τους πιο ευάλωτες ομάδες, ειδικά τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Ε, στέγαση και τροφή ε, πρόσκαιρη και ανεπαρκή σε καταβλισμούς που ε, φιλοξενούν 100.000 ανθρώπους. Εγώ έχω επισκεφθεί τη Μόρια στη Μυτιλίνη και είδα την ε, απάτη αυτή που είναι αυτά τα κοντέινερ. Τα κοντέινερ είναι ψυγεία το χειμώνα και σάουνες το καλοκαίρι. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για κατάλληλη χρήση των κονδυλίων. Όντω έχει γίνει αυτό, αλλά είναι ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο να δίνει τα χρήματα και να φτάσουν εκεί δηλαδή, αλλά να ελέγξει και τη σωστή χρήση αυτών των χρημάτων. Καταφέραμε να προχωρήσουμε στην διάσωση στη θάλασσα, αλλά τώρα πεθαίνουν εκεί στα σύνορα και η βασική προτεραιότητα είναι να σωθούν ζωές. Δεν μιλάμε για φιλοσοφίες εδώ, μιλάμε για τον τίτλο που εδώ μας αφορά, μιλάμε όχι για επίγουσα ανάγκη, μιλάμε για κατεπίγουσα ανάγκη και για αλληλεγγύη και μιλάμε για την ε, ε, κατεπίγουσα ανταπόκριση 21 και 80 είναι τα άρθρα της συνθήκης και της συνθήκης λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει ωστόσο άμεσα είναι να δεσμευτείτε ε, και όχι ε, πρόεδρε του Συμβουλίου για την Τουρκία. Πει μου μιλάτε για την Τουρκία, γιατί αυτή δεν είναι κομμάτι αυτής της συζήτησης. Εδώ ε, έχει να μιλήσει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα άλλο. Και ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Διές Μέρα, δέχεστε μπλε κάρτα. Κύριος Χόρτας, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ για την ομιλία σας και για τη λόγια σας υπέρ της ε, συμβιβαστικής λύσης. Αλλά ξέρετε ότι πολλοί που έχουν παγιδευτεί αυτή τη στιγμή κάτω από το χιόνι στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν τηρούν τις ε, δεσμεύσεις όσον αφορά τη μετεγκατάσταση. Εσείς θεωρείτε πως η κυβέρνηση ισπανική ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της όπως θα έπρεπε. Έχει, έχει δεχτεί μόνο 6% από τους πρόσφυγες που δεσμεύθηκε να υποδεχθεί στον μηχανισμό μέσω μάλλον του μηχανισμού που συμφωνήθηκε στην από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Δίαδης Δεμέρα, μάλιστα, κύριε συνάδελφε, τα λόγια μου αφορούν ε, και συμπεριλαμβάνονται στη συμβιβαστική και στην συμπόνια και αφορούν οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτά που λέω δεν έχουν να κάνουν με μια συγκεκριμένη κατάσταση. Συμφωνώ. 8.000 άνθρωποι ε, ε, προβλέπονταν εκεί σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά αυτό για το οποίο εγώ μιλάω τώρα δεν είναι, αυτό, ε, τώρα, δεν είναι αυτό που λέτε εσείς που μιλάτε με πολιτική σκοπιμότητα. Εγώ μιλώ απλά για κατεπίγουσα ανάγκη, κατεπίγουσα περίπτωση η οποία είναι ορατή και η συμπόνια ξεπερνά και υπερβαίνει οποιαδήποτε θετική ή αρνητική δράση και ενέργεια οποιασδήποτε κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ, πολύ. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσε, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, Ευρώπη όλοι έπεσε χιόνι και ανησυχούμε όλοι για τις 10.000 ε, πρόσφυγες οι οποίοι ζουν σε αυτή την παγωμένη κατάσταση. Είδαμε φοβερές εικόνες, ντρεπόμαστε, συγκινηθήκαμε, λυπόμαστε. Ενώ το χιόνι μπορεί να είναι και πηγή χαράς για κάποιους άλλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που σήμερα είναι εδώ υπεύθυνο επίτροπος γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν κάποια μέσα να διατεθούν εκεί που πρέπει. Αυτό που τελικά συνέβη είναι κάτι που φοβόμασταν, που το είχαμε ανακοινώσει. Δηλαδή υπάρχει το θέμα της μη μετεγκατάστασης. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, για τους οποίους έχει προβλεφθεί να πάνε κάπου αλλού, η γραφειοκρατία όμως, οι δύσκολες συνθήκες ζωής, οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος κάθε εβδομάδα μας λέει ότι την άλλη εβδομάδα θα βελτιωθεί η κατάσταση. Μα κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να περιμένουμε. Χρειάζεται μια ειδική ομάδα, μια task force για να λυθεί επιτέλους αυτό το θέμα. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, η κατάσταση που επικρατεί στα hot spots στην Ελλάδα είναι επικώς απαράδεκτη λόγω της υπερσυγκέντρωσης χιλιάδων προσφύγων και παράνομων μεταναστών. υπερσυγκέντρωση που οφείλεται στο ότι η τουρκία συνεχίζει να στέλνει πρόσφυγες στα νησιά του αιγαίου όπου έχουν εγκλωβιστεί 16.500 άτομα καθώς υπάρχουν μόνο 7.000 θέσεις φιλοξενίας. υπερσυγκέντρωση που οφείλεται στο γεγονός ότι το νάτο και η frontex αντί να περιορίσουν τις προσφυγικές ροές κάνουν κυριολεκτικά τον τροχονόμο. υπερσυγκέντρωση που οφείλεται στο γεγονός ότι από τους 66.400 πρόσφυγες που υποτίθεται ότι έπρεπε να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ένωσης έχουν μετεγκατασταθεί μόνο 8.000 άτομα. Υπερσυγκέντρωση που οφείλεται στο γεγονός ότι η εξέταση των αιτήσεων ασύλου χρειάζεται υπερβολικό χρόνο, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και υποσχέθηκε να στείλει εκατοντάδες ειδικού να συνδράμουν τις ελληνικές αρχές, δεν το έχει πράξει. Κύριε Στυλιανίδη, καταγγείλαμε σε όλους τους τόνους το γεγονό ότι η κυβέρνηση άφησε χιλιάδε πρόσφυγε μέσα στο χιόνι ειδικά στη μόρια τη λέσβου αλλά και στη ριτσόνα. όμω η κατάσταση στη σάμο αλλά και στη χίο όπου βρέθηκα το σαββατοκύριακο δεν είναι καλύτερη. και αυτό παρότι οι περίφημε μκο έχουν πάρει εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων. πού πήγαν λοιπόν τα λεφτά κύριε στυλιανίδη; γιατί οι μκο κάνουν πάρτι με τα λεφτά για τους πρόσφυγες. εδώ σε αυτή την αίθουσα από τον οκτώβρη έχω ζητήσει να παρέμβει η όλαφ για το ζήτημα αυτό και να γίνει έλεγχος. ακόμη περιμένω κύριε Στυλιανίδη απάντηση στην ερώτηση που υπέβαλα τον οκτώβριο για την κακοδιοίκηση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης των κονδυλίων που έχουν πάει για τους πρόσφυγες. περιμένουμε μια απάντηση. υπάρχουν ευθύνες και της κομισιόν υπάρχουν ευθύνες και της ελληνικής πλευράς η ελλάδα πλέον δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες αλλά και οι πρόσφυγες δεν μπορούν να είναι μέσα στο κρύο. ευχαριστώ. κυρία Βίξτρομ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει στα ελληνικά, κυρία Βίξτρομ. Το χιόνι συνεχίζει να πέφτει και ο πολύ βαρύς χειμώνας έχει κατακλείσει ακόμα και τον νοτιότερα τμήματα της Ευρώπης. Είναι απαράδεκτες οι συνθήκες ζωής των προσφύγων. Ευτυχώς υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες, να αναγνωρίσουν και να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα βλέπουμε τις ευρωπαϊκές ε, κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να πρέπει να αντιμετωπίσουν την καλή διαχείριση. Οι συνθήκες ε, ζωής είναι απαράδεκτες είναι απαράδεκτες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν στις όχθες μας και ζήτησαν τη φιλοξενία μας. Πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτή την κατάσταση. Βεβαίως ε, η μετεγκατάσταση αυτών των προσφύγων και όπως είχε προβλεφθεί από την Ελλάδα και την Ιταλία, δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό πρέπει να το διαπιστώσουμε. Γι' αυτό και θα πρέπει να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις και ιδέες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καλύτερα αυτή η κατάσταση. Αυτό όμως είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Άμεσα και με επίγοντα τρόπο θα πρέπει να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες αυτές της νιώτης Ευρώπης. Να τους παρέχουμε βοήθεια. Σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι ανθρωπιστική βοήθεια, κατεπίγουσα βοήθεια. Χρειάζεται συμπόνια, πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε αυτήν την τραγική κατάσταση. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε λοιπόν σήμερα. Αυτό επίγει. Σας εύχομαι κάθε καλό κύριε Επίτροπε για τις προσπάθειές σας να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Μιλούσατε εκ μέρου των φιλελευθέρων και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σπινέλη για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Διερωτώ με πόσοι τούντες άσυλο θα πρέπει να πεθάνουν από το κρύο αυτό το χειμώνα ε, στην τροπή μας μέσα. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει τη Διεθνή Αμνηστία και τη Refugee Community Leader της Μόρια. Οι μετανάστες από τα ελληνικά νησιά πρέπει να πάνε προς την υπηρετική χώρα και χωρίς να πηγαίνουν σε καταβλισμούς χωρίς ηλεκτρισμό και νερό. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας δεν προβλέπει οι παναπατρισμοί να γίνονται από τα νησιά όπως ζητήθηκε. Υπό αυτούς τους όρους και συνθήκες οι πρόσφυγες στην Ευρώπη δεν ε, πρέπει, ε, δεν πρέπει να στέλνονται στην Ελλάδα και την Ιταλία για να στεβαστούμε το Δουβλίνο. Αυτή δεν είναι μια κρίση των προσφύγων αλλά είναι μια κρίση των δικών μας πολιτικών ασύλου, μεταγκαταστάσεως, οικογενειακής επανένωσης και σεβασμού του δικαιώματος της ζωής. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, αυτό το χειμώνο, τον τόσο ψυχρό, δεν ήταν κάτι απρόβλεπτο αυτός ο χειμώνας. Με τους πρόσφυγες της Μόριας ζητώ να σταματήσουν οι απελάσεις προς την Τουρκία των πλέον ευαλώτων και να εγγυηθούμε, να δοθούν όλες οι διαδικαστικές εγγυήσεις που έχουν δικαίωμα οι διετούντες άσυλο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ, εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Φανταστείτε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τον 21ο αιώνα είμαστε και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν, που παγώνουν, τα παιδιά ε, που έχουν κρυοπαγήματα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 21ο αιώνα και εμείς φαινόμαστε αδύναμοι να τους βοηθήσουμε αποτελεσματικά. Πώς θα μπορούσαμε να αφήσουμε αυτό να συμβεί στη δική μας την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού οφείλεται στη λογική του να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, σε ετούντες άσυλο, όπως να τους αποκαλέσουμε εκτός και να τους κακομεταχειριζόμαστε και να μην έρθουν δεχόμαστε ότι υποφέρουν άνθρωποι ούτω ώστε να αποτραπεί το να έρθουν κι άλλοι. Αυτή είναι η Ευρώπη στην οποία θέλουμε να ζούμε. Αυτή είναι η Ευρώπη την οποία φανταστήκαμε όταν ήμασταν υποψήφιοι για αυτέ τι θέσει. Είναι κάτι αποδεκτό για μα, Για μένα είναι απαράδεκτο και για πολλού από εσά πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο. Αν δεν είναι αποδεκτό θα πρέπει να γίνουμε ρεαλιστέ, θα πρέπει να μεταφέρουμε τους μετανάστες από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα. Και το πρόβλημα είναι η συμφωνία της Τουρκία λόγω των περιορισμών δέχεται η Τουρκία μόνο πρόσφυγες που προέρχονται από τα νησιά. Αλλά δεν δέχεται πρόσφυγε από τα νησιά. Αλλά βάζουμε το Συμβούλιο και εμά σε δύσκολη θέση. Πιέζει η Τουρκία την Ελλάδα να μην μεταφέρει πρόσφυγες προ την υπηρετική ε, ε, Ελλάδα. Γι' αυτό έχουν κολλήσει οι άνθρωποι στα νησιά που δεν υπάρχει στέγαση και τίποτα άλλο. Και θα πρέπει να μεταγκατασταθούν, να μεταγκατασταθούν και να ξαναμεταγκατασταθούν. Μόνο 6,4% από τους 160.000 ανθρώπους έχει μεταγκατασταθεί μέχρι τώρα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Χρειαζόμαστε δράση από πλευράς κρατών μελών. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχουμε τη Σερβία, έχουμε τη Μακεδονία, έχουμε τη Βουλγαρία, όπου εκεί πρέπει να αυξήσουμε τις ε, δυνατότητες υποδοχής και στέγασης. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να σταματήσουμε να Υπόκρινόμαθα ότι θα σταματήσει να φεύγει ο κόσμο από σύγκρουση, δίωξη και πόλεμο, εάν κάνουμε την κατάσταση εδώ φρικτή για αυτού. Αυτό δεν θα συμβεί. Πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα και τελικά να δώσουμε κάποια αξιοπρέπεια στου ανθρώπου αυτού, αλλά και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πέρασε ένας άλλος χρόνος με ελάχιστη πρόοδο και βελτίωση. Μιλάμε για προσωρινές ε, λύσεις για κάποια προβλήματα τα οποία φαίνεται να γίνονται μόνιμα. Στην ε, Σουηδία οι σοσιαλδημοκράτες μιλούν πάντα για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται και ζούνε από το να προσπαθούμε να τους προσελκύσουμε και να τους βοηθήσουμε στις δικές μας χώρες. Να προλάβουμε δηλαδή το πρόβλημα πριν να μεγαλώσει και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ήδη από το 2011 έχει ξεκινήσει η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Εμείς στην Σουηδία αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε σκηνές και παραπήγματα γιατί είχαμε δεχτεί ένα υπερβολικά υψηλό αριθμό προσφύγων. Είχαμε δηλαδή δεχτεί στη χώρα μας χώρες που δεν μπορούσαμε να, τις, ε, να τους ε, βοηθήσουμε. Είμαστε η χώρα εξάλλου που δέχτηκε πέρσι το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ε, ανακάτοικο. Πώς λοιπόν θα συνεχίσουμε με αυτές τους διπλούς κανονισμούς και πότε θα τηρήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπρουά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτίμηση στους αλλοδαπούς. Αυτό είναι κάτι το σκανδαλώδες. 120, 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με άθλιες συνθήκες και κανείς ε, σήμερα πιο ευνοϊκά αντιμετωπίζεται αν είναι μετανάστης ή πρόσφυγας από το να είναι φτωχός Ευρωπαίος. Σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε με την ίδια επίοικια και συμπόνια τους ε, άστιγους ε, Ευρωπαίους. Έχουμε δημιουργήσει μια ιεραρχία στη φτώχεια και στη μιζέρια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δείξουμε κοινή λογική στη χώρα μου. Κάποιοι πολιτικοί, όπως η Δήμαρχος του Παρισιού, έχει δημιουργήσει συνθήκες φιλοξενίας για μετανάστες και πρόσφυγες και αφήνει με αδιαφορία τους άστεγους στα πεζοδρόμια και στους δρόμους πρέπει πρώτα να σκεφτούμε τους δικούς μας ανθρώπους και μετά τους αλλοδαπούς. Ευχαριστώ πολύ κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό. Τρόπε, Γενάρη μήνα θα κάνετε προσαρμογή όπως λέτε για το χειμώνα και σήμερα στη Λέσβο προτείνατε πάλι σκηνέ. Με δήλωσή της ΔΕΗ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δηλώνει μάλιστα ικανοποιημένη. Ισχυρίζεται αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία ότι 57.000 είναι στεγασμένοι και με θέρμανση. Ομολογεί ότι οι υπόλοιποι δηλαδή 6.000 ξεπαγιάζουν με κίνδυνο ζωής πρόκειται για απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας που τους καταδίκασε σε διπλό εγκλωβισμό σε απερίγραπτες συνθήκες περιμένοντας βασανιστικά άσυλο ενώ οι μκο λιμένονται όλα αυτά τα κονδύλια και κανοναρχούν στα κάμπ. αυτά όλα είναι αποτέλεσμα της κοινής απόφασης ευρωπαϊκής ένωσης και όλων των κυβερνήσεων όχι μόνο του βίζεγκραντ να κλείσετε τα σύνορα να χτίσετε τείχη με καταστολή απελάσεις ευρωσυνοριοφυλακή άμεσα τώρα να μετακινηθούν από τα νησιά οι διπλοεγκλωβισμένοι να μεταφερθούν στις χώρες τελικού προορισμού τους. επίγουσα ανάγκη κανένας πρόσφυγας και μετανάστης σε σκηνή κανένας χωρίς θέρμανση ρεύμα νερό κατάλληλη για το χειμώνα σύτηση ένδυση κρατική περίθαλψη έξω από τα κέντρα η καμιά δημιουργία κέντρου κράτησης και κάτω τα χέρια των φασιστών της χρυσής αυγής από τα προσφυγόπουλα και το δικαίωμά του στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, δεν άκουσα το όνομά μου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία μετά την επανεκλογή σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το πρόβλημα που συζητάμε είναι πάντα επίκαιρο και δυστυχώς οξύνεται γιατί τα προβλήματα αυξάνονται. στην ελλάδα στη χώρα μου ξέρετε ότι ο στόχος της μετεγκατάστασης μέχρι το σεπτέμβριο του δύο πρέπει να είναι δύο με τρεις χιλιάδες το μήνα. μέχρι σήμερα έχουν μετεγκαταστηθεί μόνο επτά χιλιάδες άτομα κάτι που σημαίνει ότι ο θεσμός έχει αποτύχει. επίσης απειλείται το λέω εντός εισαγωγικών το ρήμα επανέναρξη των μεταφορών σταδιακά από το μάρτιο του 2017 δηλαδή επανενεργοποίηση της συνθήκης του, δουβλίνου που όπως ξέρετε από το 2011 είχε ανασταλεί κάτι το οποίο βοήθησε τη χώρα εν μέρη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. επίσης σύμφωνα με τη συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας πρέπει να γνωρίζετε με επίσημα στοιχεία ότι έχουμε καθημερινές αφήξεις αλλοδαπών 150 περίπου άτομα δηλαδή περίπου 4.000 το μήνα. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα νησιά έχουν συγκεντρωθεί δεκαέξι άνθρωποι και παρά το γεγονός ότι το ελληνική πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί δεν έχει μπορέσει να διαχειριστεί στην επάρκεια το πρόβλημα γνωρίζετε όλοι ότι ο ελληνικός λαός έχει δείξει δείγματα θαυμαστού ανθρωπιστικού έργου προς τους ανθρώπους αυτούς που ποτέ δεν αντιμετώπισε ως αριθμούς αλλά ως ανθρώπους. το πρόβλημα είναι όμως οξύ και πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να βοηθήσει το λέω γιατί ξέρετε όλοι σας ότι μία και μόνη χώρα ένα και μόνο κράτος δεν μπορεί να το καταφέρει καταφέρει και αν η ελλάδα αποτύχει στη διαχείριση αυτού του πολύ σημαντικού προβλήματος θα έχει αποτύχει όλη η ευρωπαϊκή ένωση. σας ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τις τελευταίες μέρες οι τηλεοράσεις ορισμένων από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούν για κύμα ψύχου στις χώρες τους. Μιλούν για ξεσπάσματα γρήπης και για ε, κατάσταση επίγουσα. Όμως εκεί που υπάρχει όντως επίγουσα ανάγκη είναι στα Βαλκάνια, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στην Τσεχική Δημοκρατία, σε διάφορα σημεία στη Σερβία, όπου χιλιάδες και χιλιάδων ε, πρόσφυγες περνούν, περάσαν τα Χριστούγεννα σε πραγματικό κύμα ψύχους, ε, σωματικό και ηθικό κύμα ψύχους, εγκαταλελειμμένοι από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ένωσης που δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους ε, ε, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν στα σύνορά μας. Πρόκειται για μια επίγουσα βοήθεια, τρόφιμα, ε, στέγη, φάρμακα, νομική συμβουλή, βοήθεια βοήθεια κάθε είδου, Αλλά πρέπει επίση να ξεκινήσει ένα μέσο και μακροπρόθεσμο σχέδιο, αυτό το winterization plan, το, η προσαρμογή σε χειμερινές συνθήκε δηλαδή και πρέπει ε, τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πια αυτήν τη, τη, τη, δέσμευση και να ανταποκριθούν σε αυτή. Κύριε Κυρέρο, δέχεστε ερώτηση από την κυρία Σόιντροβα. Παρακαλώ. Uh, Ήθελα να ρωτήσω, πού πήρατε τις πληροφορίες που μόλις αναφέρατε. Αληθεύει ότι κάνει πολύ κρύο στην τσεχική δημοκρατία. Πράγματι, έχουμε άστεγους στην τσεχική δημοκρατία, οι οποίοι δεν έχουν πουθενά να μείνουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν ελεύθερες θέσεις σε καταβλισμούς, σε χώρους για ετούντες άσυλο, σε σπίτια για ετούντες άσυλο δεν αληθεύει ότι πεθαίνουν ετούντες άσυλο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ετούντες άσυλο εξεπλάγην από αυτά που μόλις μας είπατε. Κοιτάξτε, είδα τους πρόσφυγες, αλλά ε, η Διεθνής Οργάνωση Προσφύγων, η ΑΚΝΟΥΡ, η Διεθνής Αμνηστία και τα στοιχεία της Κομισιόν που γνωρίζει ότι πολλά μέρη στην Ένωση συμπεριλαμβανομένων κάποιων ε, ε, σημείων στην Τσεχική Δημοκρατία υποφέρουν από αυτήν την κατάσταση. Εγώ δεν είμαι κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας. Άλλες χώρες έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από την Τσεχία και δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους. Και η δικιά μου χώρα είναι μεταξύ αυτών. Γιούρε, λοιπόν, Γιούρεκ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν την ανθρωπιστική κρίση. Εκεί που ξεκινάει αυτή η καταστροφή θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για πολιτική. Στηρίζω όλους αυτούς που λένε ότι τα κονδύλια που δίνονται για βοήθεια προς αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής θα πρέπει να παρακολουθούνται, θα πρέπει πραγματικά να διοχετεύονται στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Όταν συμβαίνει μια τέτοια ανθρωπιστική κρίση θα πρέπει να σταματάμε την πολιτική. Είμαστε υπεύθυνοι πολιτικοί και με μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε ποιος δεν έπαιξε σωστά το ρόλο του και που δεν έγινε σωστά η διαχείριση. Σήμερα υπάρχει μια μαφία ε, παράνομων ε, μεταναστών και πραγματικά ε, αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω μία μαφία η οποία συνεχίζει να δραστηριοποιείται. Δεν πήραμε απολύτως κανένα, κανένα μέτρο και δεν έχουμε κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των απλών με προσφύγων και των μεταναστών. Δεν υπάρχει εντολή για να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας. Όλοι αυτοί οι μαφιόζοι έχουν ανοίξει τις πόρτες και εδώ και χρόνια κινητοποιούν γη και ουρανό για να κερδοσκοπήσουν. Συνεχίζουν το εμπόριό τους Ο κύριος Γκέρενς, ο Επίτροπος Τηλιανίδης, μας έκανε πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και με επίγοντα τρόπο να αναλάβουμε μία δράση να σταματήσουμε να ψάχνουμε τους υπεύθυνους για τα προβλήματα και την έλλειψη ε, αποτελεσματικής δράσης τα τελευταία χρόνια και να αρχίσουμε πραγματικά να παρέχουμε την κατεπίγουσα βοήθεια που χρειάζεται. Βεβαίως και θα πρέπει να κατανεμηθούν τα βάρη μεταξύ των 28 και να μην αφήσουμε την Ελλάδα και την Ιταλία μόνες τους, χώρες με σοβαρές δυσκολίες, ακόμα και πριν την μαζική προσέλευση προσφύγων και μεταναστών. Αντί να επιτεθούμε κατά της Επιτροπής, ας επιτεθούμε προς κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες για λόγους λακιστικούς, δημαγωγικούς, αρνούνται να βοηθήσουν, αρνούνται να αναλάβουν ένα τμήμα αυτού του βάρους. Εάν στηρίξουμε τον Επίτροπο Στυλιανίδη και καταφέρει να κατανείμει αυτά τα κονδύλια έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι κάποια κράτη-μέλη αρνούνται και με ντροπιαστικό τρόπο αρνούνται να δώσουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες στην Επιτροπή και επιμένουν με θράσος να επιτίθενται κατά της Επιτροπής για δίθεν έλλειψη δράσης. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπιόρκ. Η κατάσταση αυτό το χειμώνα είναι απάνθρωπη, παγώνει ο κόσμος από το κρύο, παγώνουν σε καταβλισμούς το 2017. Όχι γιατί πρέπει, εμείς δημιουργήσαμε αυτή την κατάσταση. Είναι απάνθρωπες οι πολιτικές αποφάσεις που λάβαμε, λανθασμένες. Τι είναι αυτή η Ευρώπη που έχουμε, η μαύρη τρύπα της αδιαφορίας είναι. Κλείσαμε τα σύνορα, ε, χιλιάδες πρόσφυγες βρίσκονται στην Ελλάδα, οι υπόλοιποι στα Δυτικά Βαλκάνια. Και πρέπει να στέλνουμε και ανθρώπους, όταν να στείλουμε κάποιους να ελέγχουν τα σύνορα, το κάνουμε. Εάν είναι να βοηθήσουμε του πρόσφυγε, κανεί δεν κάνει τίποτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα ακούσαμε αυτά. Αυτά που γίνονται δεν είναι αρκετά. Έχουμε μια καταστροφή που συμβαίνει τώρα. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη-μέλη εκείνα να κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από εκείνους που δεν θέλουν να κάνουν κάτι. Θα πρέπει εκείνοι που να μπορούν να συμμετάσχουν να συμμετάσχουν. Θέλουμε να γίνει ε, κατεπίγουσα κατάσταση. Θέλουμε να κλείσουμε τους καταβλισμούς στα νησιά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρζεντίνη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 18 μήνυ λεωφορεία τέσσερις γεννήτριες, 300, 300 ε, ράντζα, ε, στρώματα, 200 σέτες εντόνια και ε, κάποιες εκατοντάδες αντλίες νερού. Αυτά δώσαμε στην Ελλάδα για να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα των προσφύγων. Αυτό είναι επίγουσα βοήθεια που ήρθε από την Ολλανδία και άλλες χώρες. Επίγουσα βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση για την οποία εν μέρει είμαστε υπεύθυνοι γιατί αρνηθήκαμε να πάρουμε πρόσφυγες από την Ελλάδα και την Ιταλία. 10.000 πρόσφυγες τους υποσχέθηκαν ότι θα επανακατασταθούν αλλού στην Ολλανδία. Ας πούμε η Ολλανδία κλείνει τα κέντρα επαναγκατάστασης. Ε, ε, και μάλιστα θα σκεφτόταν κανείς ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση αυτή των προσφύγων με στα χιόνια, τις φωτογραφίες που είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πραγματικά σοκαριστικό να βλέπεις μια τέτοια κατάσταση. Δεν κάνουμε απολύτω τίποτα. Ο κύριος Συναδεινός. Πολλοί εντός και εκτός κοινοβουλίου φορώντας το μανδύα του ανθρωπιστή με πολιτική ταυτότητα και άποψη που θέλουν να επιβάλλουν μιλάνε για το δράμα προσφύγων και λαθρομεταναστών. δηλώνουν ανθρωπιστέ, αλλά στην πραγματικότητα ξεχνάνε να είναι άνθρωποι. στην ευρώπη και ειδικά στη χτυπημένη από τα μνημόνια ελλάδα υπάρχουν άνεργοι που αδυνατούν να επιβιώσουν οικογένειε χωρί στέγη ρεύμα τρόφιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. συνάνθρωποι και ομοεθνεί μα που προσβλέπουν στον ανθρωπισμό όλων μα το δράμα όλων αυτών δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε ή να το τοποθετούμε σε δεύτερη μοίρα. Ασφαλώ και οφείλουμε ω άνθρωποι και χριστιανοί να βοηθήσουμε του πρόσφυγε. Κανένα όμω πολιτικό και καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να ρίχνει το βάρο τη αποκλειστικά στου λαθρομετανάστε και να αδιαφορεί για τα προβλήματα των ελλήνων και των ευρωπαίων γενικότερα. αν εμεί εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μα, τότε ηθικά και νομοτελειακά δεν έχουμε λόγο πολιτική ύπαρξη να υπενθυμίσω σε όλους εσάς ανθρωπιστές και μη ότι έχετε βήμα και λόγο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διότι σας εξέλεξαν οι συμπολίτες μας και όχι οι λαθρομετανάστες. ευχαριστώ. Υπάρχει μπλε κάρτα. Τη δέχεστε, κύριε Συνοδυνέ. Κύριε Συνοδυνέ, δέχεστε την μπλε κάρτα, κύριε Συνοδυνέ. Ναι. ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που είπατε. Από τη μία μεριά βάζετε τους πρόσφυγες και από την άλλη τους μετανάστες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι μεν και οι δε, οι οποίοι πρέπει να τύχουν ανθρώπινης μεταχείρισης. Μπορεί να συμφωνούσα σε αυτό που λέτε, εάν υπήρχε κάποιο διαχωρισμό εδώ και τόσο καιρό που συζητάμε σε αυτό το κοινοβούλιο για του πρόσφυγε και του λαθρομετανάστε. σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο άλλο είναι το ημέν και άλλο είναι η δε. ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Χιμένες για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε για την ε, ε, συμπόνιασε σε μια τόσα πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην Νότια Ευρώπη. Με λυπή η ευρωπαϊκή απάθεια όταν βλέπουμε ε, θανάτους κάτω από αυτό το κύμα ψύχους. Ε, βλέπουμε τα κορμάκια των παιδιών. Βλέπουμε όμως με θλίψη και σφίξιμο καρδιές ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Πέρυσι πήγα στην Λέσβος και στη Λέσβο και στην Αθήνα. Πήγα στην Μόρια. Είδατε πόσο ζέστη έκανε τώρα αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ε, υποφέρουν σε αυτές τις ίδιες σκηνέ, σε αυτό το φρικτό κρύο. Η κατάσταση είναι δραματική και γι' αυτό και θα πρέπει να είναι δραματική η αντίδρασή μας ώστε να μην ε, πεθάνουν παιδάκια από ιούς και γρήπες. Πρέπει επιγόντως να βοηθήσουμε την Ευρώπη. Χτες ε, ζέστη, καύσωνας, σήμερα κρύο. Ας απλοποιήσουμε το σύστημα ασύλου ώστε να περάσουν νόμιμα και οι άνθρωποι στην Ευρώπη ώστε να μην χρειάζεται να εξαρτώνται από τα χέρια των ε, ασυνείδητων ε, ε, διακινητών οι, επίσης οι άνθρωποι, να, να, οι, οι χώρες της Ένωσης να ανοίξουν τα σύνορά τους ώστε να μην είναι πια μια ποντικοπαγίδα η Ελλάδα ο κόσμος να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους μη ε, συνοδευόμενους ανήλικους γιατί κανένα παιδί δεν μπορεί να ζει όχι μόνο μακριά από το σπίτι του αλλά και κρύο, κρύο μέσα στην ψυχούλα του. Ευχαριστώ. Ο um, Πρόεδρε. Εγώ με την Επιτροπή Ανάπτυξης έχω παρακολουθήσει αυτές τις τραγικές καταστάσεις όπου άνθρωποι υποφέρουν από το κρύο, παθαίνουν υποθερμία, ή κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ ανησυχητική και δεν είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο είναι μεμονωμένο. Υπάρχει τέτοια κατάσταση σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Υπάρχει και στους καταβλισμούς ε, της Ιορδανίας και αλλού στον κόσμο, αλλά δεν είναι δυνατόν το 2017 να πεθαίνουν στην καρδιά της Ευρώπης πρόσφυγες από το κρύο. Και αυτό που θα ήθελα να πω στην ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συζητήσαμε το θέμα αυτό της ε, μετεγκατάστασης και ξέρουμε ότι δουλεύει πολύ σκληρά η Επιτροπή. Γι' αυτό ξέρουμε κύριε Επίτροπε ότι δουλεύετε σκληρά. Κανείς δεν αμφισβητεί τις προσπάθειές σας. Αυτό όμως που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω σε αυτήν την τόσο επίγουσα κατάσταση. Εμείς ε, στη συζήτηση που κάναμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί να γίνουν κάποια παραπάνω πράγματα. Πείτε μας ποια κατά την άποψή σας μπορούν να είναι αυτά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάκοψης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η κατάσταση στα ελληνικά νησιά είναι πέραν της ε, δραματικής. Αυτό που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η πολιτική μας απέτυχε. Εμείς, η δράση μας απέτυχε. Δεν ξέρουμε ακριβώς ε, πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Βλέπουμε τις εποχές να εναλλάσσονται μετά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ο χειμώνας και εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές. Η κατάσταση στη Σερβία είναι δραματική. Στο κέντρο του, της πόλης του Βελιγραδιού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, προσφύγων και πρέπει να βοηθήσουμε τη Σερβία, πρέπει να βοηθήσουμε την πόλη του Βελιγραδίου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να είμαστε επίσης πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το άνοιγμα του δρόμου της διαδρομής των Βαλκανίων. Η κατάσταση σήμερα για τα Βαλκάνια δεν είναι καθόλου καλή και αυτό συνεχίζει να είναι ανησυχητικό. Υπάρχουν σοβαρές εντάσεις οι οποίες αυξάνονται και οι πρόσφυγες, η κατάστασή τους σήμερα εντείνουν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρυσόγονος έχει το λόγο. Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελεί μια καλή ευκαιρία να δείξουμε περισσότερη αλληλεγγύη. οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές όπως η νησιωτική ελλάδα δοκίμασαν τις αντοχές των κρατικών μηχανισμών αλλά και των προσφύγων. είναι αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να επιβεβαιώσει την υποστήριξή της με στόχο την καταλληλότερη φροντίδα προσφύγων και μεταναστών. ήδη τα στοιχεία δείχνουν πω η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών λαμβάνει κατάλληλη φροντίδα με υλική υποστήριξη αλλά και με επιπλέον προσωπικό. Καθώ όμω οι καιρικέ συνθήκε έφτασαν τον ελληνικό κρατικό μηχανισμό στα ακραία του όρια θα πρέπει να αποφασίσουμε το συντομότερο δυνατό την παροχή επιπλέον βοήθεια στι περιοχέ που επλήγησαν από την κακοκαιρία όπω πράττουμε σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ευχαριστώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 20 Μαρτίου του 2016 όταν άρχισε να ισχύει η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία η Ελλάδα έπαψε να είναι χώρα διέλευσης αλλά και άρχισε να είναι φύλακα φύλακας όλων αυτών των χιλιάδων προσφύγων. Η Ελλάδα λοιπόν ε, δέχτηκε και 200 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Μέσο Επίγουσες Ανάγκης για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ευθύνες της, να μετατρέψει δηλαδή τους προσωρινούς καταβλισμούς σε κάτι μόνιμο. Τι έκανε η κυβέρνηση της Ελλάδας, έχει χάσει ο κύριος Τσίπρας τον έλεγχο της διοίκησης γιατί με 200 εκατομμύρια πολλά μπορούσαν να γίνουν ε, με βάση βέβαια τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις της το ποσό των 200 εκατομμυρίων στο οποίο αναφερθήκατε είναι πάρα πολύ μικρό αν αναλογιστούμε ποιο είναι ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στο ελληνικό έδαφος που είναι πάνω από 60.000 και ποιε είναι οι αντικειμενικές δυσχέρειες εν ώψη και των γεωγραφικών συνθήκων. Μικρά νησιά, υπερφορτωμένα, Συνεπώ, δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό. Δεν λέω ότι όλα γίνονται τέλεια αλλά η ευρώπη πρέπει να βοηθήσει περισσότερο. Thank you. Ο κύριος Μπούντα. Εξ ονόματος του Ντάνιελ Μπούντα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η μετανάστευση έγινε μια πραγματική οδυνηρή πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε αποτελεσματικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να χειριστούμε το φαινόμενο. Παρά το ότι βρισκόμαστε στο χώρο Σέγγεν, τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να διασφαλίσουν τα σύνορα. Σύμφωνα με τη Frontex, το 2015 πάνω από ένα 83 εκατομμύρια διελεύσεις, παράνομες διελεύσεις είχαμε των συνόρων και η αριθμή είναι πολύ ψηλότερη το 2016. Όλα αυτά τα άτομα είτε είναι οικονομικοί μετανάστες, είτε είναι μετανάστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις βόμβες, αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση σήμερα. Προερχόμενοι από ερημικές περιοχές, Μόλι φτάσουν εδώ, δεν πρέπει να πολεμήσουν μόνο τι κοινωνικέ συνθήκε, αλλά να καταπολεμήσουν και τι καιρικέ συνθήκε, οι οποίε φαίνεται να είναι σκληρότερε φέτο από ότι οποιοδήποτε προηγούμενο έτο. Και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι συνθήκε ακόμα και από του ντόπιου πληθυσμού. Επεσκέφθηκα το καλέ, τον καταβλισμό του καλέ πριν κλείσει. Ήταν ένα μέρο που σίγουρα θέλεις να λησμονήσεις ότι υπήρξε. Ένα μέρος που το λησμόνησε ο Θεός, μαρτυρίου και έδειχνε την αδυναμία να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Σήμερα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη έναντι εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όμως, ας μην λησμονούμε κάτι. Εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορούμε να έχουμε μόνο προσωρινές λύσεις. Η τελική λύση έγκυται εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, στις χώρες αυτών των ανθρώπων, όπου ασφαλείς περιοχές θα πρέπει να δημιουργηθούν για να μπορούν να διαμείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα. Η κυρία Βαλενσιάνο έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω αρκετή εμπιστοσύνη στον κύριο Επίτροπο και νομίζω ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ε, δίνει πολλές ελπίδες η Προεδρία της Μάλτας γιατί πιστεύω πως έχει ιδιαίτερη ευαισθησία ε, απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα. Το είπαν όλοι μας οι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι έχουμε κατασκευάσει ένα μεγάλο ανθρώπινο και νομικό λίμπο για χιλιάδες ε, κόσμου και κάποιες φορές αυτό το λίμπο παγώνει και φτάνει ή και άλλες φορές φτάνει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, σε καύσωνα. Και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνουμε κάτι στη δικιά μας επικράτεια ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε στα, Ευρωπα... στα ελληνικά νησιά όλο αυτόν τον κόσμο που αυτή τη στιγμή έχει παγώσει. Όπως είπαμε πρόκειται για μια παγίδα, μια βοντικοπαγίδα για πολλά παιδιά. Ε, ανήλικα που χρειάζονται διεθνή προστασία. Ε, αισθάνονται προκαταλελειμμένοι και είμαστε υπεύθυνοι, σαφώ και είμαστε υπεύθυνοι για τι πολιτικέ αποφάσει και για την ανεπάρκεια της ε, διαχείρισης. Και στρέφομαι στην ε, ε, Προεδρία της Μάλτας που θα πρέπει να επιμείνει στο Συμβούλιο, θα πρέπει να επιμείνει απέναντι στους Πρωθυπουργούς όσον αφορά την επίγουσα ανάγκη να δράσουν, ώστε αυτή η συζήτηση μια μέρα των ημερών να γίνει συζήτηση της ελπίδας και όχι της απελπισίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουλευτή. Και τώρα η κυρία Έλλη Σλάιν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, λίγες μέρες πριν είδαμε ένα βίντεο που γύρισε ένα τον άσυλο στο καταβλισμό τη Μόρια στη Λέσβο. Εκατοντάδε άνθρωποι ε, ε, ήταν υποχρεωμένοι να κοιμούνται σε σκηνέ που δεν είχαν θέρμανση, κάτω από τα χιόνια, δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν υπήρχαν κουβέρτε. Τα μέσα που εσεί ανακοινώσατε δεν αρκούν εφόσον είναι τέτοια κατάσταση. Σα καλώ να το αυξήσετε και να ελέγξετε πώ χρησιμοποιούνται τα κονδύλια τη Κομισιόν ώστε να εξασφαλιστούν ανθρώπινε συνθήκε διαβίωση, Οι γιατροί χωρί σύνορα και άλλες ΜΚΟ καταγγέλουν πολύ σοβαρές καταστάσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στη Σερβία όπου έχει μείον 20 βαθμούς και άνθρωποι είναι τελείως εγκαταλελειμμένοι. Ο ΙΕ θέλει να μετακινήσει 15.000 κόσμο από τα νησιά στην πυρωτική Ελλάδα για να υπάρξει καλύτερη στέγαση οι δε τοποθετήσεις αυτές είναι σταθερές μόνο για το 12%. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό το μηχανισμό που ήδη είχε ενεργοποιηθεί από το 2015. Δεν είναι αποδεκτό να μένει στο κρύο κανένας, κύριε Επίτροπε. Τι θα κάνετε ώστε να στεγαστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σλάιν και τώρα η κυρία Μακάβαν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι. Και ξέρουμε, οι ΜΚΟ μα λένε ότι είναι χάλια συνθήκες στέγας αυτών των ανθρώπων. Χιλιάδες έχουν αποκλειστεί στη Βαλκανική Οδό και πολλά παιδιά. 300 συνόδευτα παιδιά ε, ζουν σε άθε συνθήκες στο Βελιγράδι. Πρέπει κατεπηγόντως να γίνει κάτι. Ένα Βαλενσιάνο αναφέρθηκε στο κενό αυτό, τον κενό χώρο, το λίμπο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων, να γίνουν όσο πιο άνετοι γίνονται οι συνθήκες διαβίωσης. Ένας τρόπος να το πετύχουμε είναι να έχουν κάποιο σύστημα με δελτία ε, για να παίρνουν τρόφιμα αντί να περιμένουν να πάρουν σούπα, θα μπορούν να τους δώσουμε ε, μετρητά να αγοράσουν από ντόπιου ε, πολιτές τρόφιμα. Έχει επιτευχθεί πρόοδος αυτό. Και τι γίνεται με την εκπαίδευση των παιδιών, με την παιδεία των παιδιών. Είναι προτεραιότητα αυτό για σας κύριε Επίτροπε. Θα θέλαμε ενημέρωση γι' αυτό. Από την Προεδρία της Μάλτα ξέρουμε ότι κάνετε ό,τι μπορείτε. Ξέρουμε ότι δεν, είναι, δεν θέλω να επικρίνω την Ελλάδα, ούτε η χώρα μου έκανε κάτι παρόμοιο καν από αυτά που έκανε η Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολε καταστάσει και για την Ελλάδα, πολύ δύσκολη. Πρέπει όλοι να ενωθούμε και να αντιμετωπίσουμε κατεπίγους ανάγκη. Και βέβαια έχουμε και τα μεγάλα θέματα διαμόρφωση πολιτική, τα οποία θα πρέπει να επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Πάμε στη διαδικασία Catch the Υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Η κυρία Μιχέλα Σόιτροβα έχει το λόγο πρώτη. Σας ευχαριστώ, επίτροπε συνάδελφοι. Πάλι πιαστήκαμε στον ύπνο. Το 2014, το 2015 μας εξέπληξε το μεταναστευτικό κύμα ε, των ε, και πάλι τώρα μας εκπλήσει ότι στα hot spots στα ελληνικά νησιά επικρατούν άθλιες συνθήκες για τον κόσμο που χρειάζεται βοήθεια. Κανένας δεν περίμενε τέτοιες καιρικέ συνθήκες. Βλέπουμε πως η Ευρώπη είναι απροετοίμαστη. Δεν είμαστε σε θέση να προβλέπουμε τέτοιες καταστάσεις που μπορεί ωστόσο να συμβούν. Οφείλουμε να συνεργαστούμε. Ένα μόνο κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, τέτοιες δυσκολίες. Και με χαρά από τον Επίτροπο πως υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. Ε, το ερώτημά μου είναι όμως τι θα έπρεπε να έχουμε ήδη κάνει ώστε να μην βρεθούμε σε τόσο άσχημη κατάσταση κάτι ξεχάσαμε. Κάτι σίγουρα ξεχάσαμε. Τι ακριβώς ήταν αυτό. Έπρεπε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόνο στο Βελιγράδι χιλιάδες άνθρωποι έχουν μπλοκαριστεί στο κρύο και κινδυνεύουν να πεθάνουν. Τόσε οικογένειε, πάρα πολλά παιδιά προσπαθούν αυτέ τι μέρε ε, να εξεγαστούν σε εγκαταλειμμένα κτίρια. Ζητούμε ανθρωπιστική προστασία από την Ευρώπη και εμεί τελικά σημειώνουμε, ε, σηκώνουμε τείχου και σειρματόπλεγμα για να εμποδίσουμε τη ροή των απελπισμένων. Απαντά μην εφαρμόζοντα τι διεθνεί νομοθεσίε που εγγυώνται το δικαίωμα στην ανθρωπιστική προστασία. Αυτή η Ευρώπη που τιμωρεί εκείνον που ε, δεν δημιουργεί κοινού παραβίαση ανθρώπινα δικαιώματα, δεν σέβεται του κανόνε. Όπω στη χώρα μου, που εδώ και χρόνια προσπαθεί να σώζει τη ζωή των ανθρώπων στη θάλασσα η χώρα μου. Λοιπόν, γυναίκε και παιδιά ε, καταδικάζονται σε θάνατο. Αυτή δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Ήρθε η στιγμή να δράσουμε. Χρειάζεται κινητοποίηση. Να βοηθήσουμε αμέσω αυτά τα πολλά άτομα λιώνοντας τον κόμβο της κοινική αντιμετώπισης που δείχνουν κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπούτο. Και τώρα στον κύριο Λόπες Αγιλάρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτροπή Προεδρία της Μάλτας, όταν στο τέλος κάθε εξαμήνου η Προεδρία συγκεντρώνεται στο Συμβούλιο και το κάνει ώστε οι αρχικοί κρατών και κοινοβουλίων να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Όμως όταν παρακολουθείτε εδώ, έρχεστε όχι μόνο για να συζητήσετε μαζί μας, αλλά και για να ακούσετε. Οι εκπρόσωποι των, των, ανθρω... των λαών μας έχει εξαγριωθεί ε, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, απέναντι στην παγωνιά και απέναντι σε αυτή την άθλια κατάσταση των ε, προσφύγων προσφύγων. Μπορείτε να στηρίξετε τον ευρωπαϊσμό σας ε, αφού έχω ζήσει σε πρώτη γραμμή τη δραματική κατάσταση της ε, μεταναστευτικής ε, ροής που την αποκαλέσαμε κακώς προσφυγική κρίση. Πρόκειται για μια ατελείωτη κρίση που από το 2008 την έχουμε διαχειριστεί χείριστα ε, Πώ μπορείτε να εξηγήσετε και να απαιτήσετε από τι κυβερνήσεις να τηρήσουν τις δεσμεύσει όσον αφορά την επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση και, να μην, και επίσης να, ε, να, ε, να ξεπαγώσουν το πακέτο για το άσυλο, το πακέτο το θεωρήσεων ώστε να δημιουργηθούν νόμιμες οδοί ώστε να φτάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι για μια τέτοια κατάσταση ανθρωπιστικές βίζες, ανθρωπιστική διάδρομη. Προεδρία της Μάλτας, Μιλήστε με τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο, με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση που να μπορεί να αποκαλείται ανθρωπιστική. Δεν είναι κρίση ανθρωπιστική, είναι ε, ε, προσφυγική, είναι ανθρωπιστική η κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Σεσίλια Κέγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ζητούμε μία παρέμβαση κατεπηγόντω. Ζητούμε την κατεπίγουσα αυτή παρέμβαση για να εξασφαλίσουμε ενίσχυση βοηθεία για χιλιάδε ετούντε άσυλο και μετανάστε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίε λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, με χιόνι και παγωνιά στην Ευρώπη. και όμως όλα θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί. Θα μπορούσαμε να δράσουμε εγκαίρως αλλά παρέμειναν ακόμα με αυτή την προσέγγιση τη αντιμετώπιση κατεπίγουσα ανάγκη. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό για να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε προγράμματα μέσω μακροπρόθεσμα. Ε, χρειαζόμαστε με αυτό το νέο εργαλείο της ανθρωπιστικής βοήθειας επί ευρωπαϊκού εδάφους να δράσουμε αποτελεσματικά. Ε, δεν πρέπει να ανεχτούμε καθυστερήσεις, πρέπει να είμαστε παρόντες εκεί που αφέρουν οι άνθρωποι, εκεί που άνθρωποι έχουν ανάγκη χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να ενεργοποιηθεί τάχιστα, να κινητοποιηθεί με τα κράτη-μέλη και κυρίω να ξεπεράσει του εγωισμού των κρατών μελών. Πρέπει να σώσουμε ζωέ. Όχι, δεν θέλουμε να οικοδομήσουμε τύχη. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να είναι ευέλικτη. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, Jolly κυρία Τζούλι Ward έχει το λόγο. Συνάδελφοι, κάποιοι ασχολούνται με κάποιες συμφωνίες δίνοντας την ψήφο τους αυτόν που θα δώσει τα περισσότερα και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι δίνουμε μια τελείως λαθασμένη εικόνα όσον αφορά το Brexit και άνθρωποι την ίδια ώρα παγώνουν στους δρόμους Ευρώπης. Πρόκειται για, μετανα... για πρόσφυγες, για ανθρώπους που ζητούν άσυλο, οι οποίοι έχουν διαφύγει τις πατρίδες τους όπου επικρατεί ε, πόλεμος. Πρόκειται για ανθρώπους που φτάνουν ε, στην ε, Ελλάδα, στα νησιά, σε καταβλισμούς, στους οποίους πρόχνουν προς τα πίσω εχθρικές κυβερνήσεις στα Βαλκάνια βλέπουμε ότι η στάση των κυβερνήσεών μας είναι αμήλικτη και υπάρχουν ευτυχώς οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που στηρίζουν και βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ οι κυβερνήσεις μας έπρεπε να στηρίξουν και να βοηθήσουν, δεν το έχουν κάνουν. Και αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να στηρίξουμε σε προσωπικό επίπεδο με την δράση μας ε, αλλά και με την κατεπίγουσα βοήθεια που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Όλοι οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να δείξουν συμπόνια. Και ευχαριστώ πολύ αυτούς που το κάνουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί από τη δική μου επικράτεια στην ε, Βορειοδυτική Αγγλία απλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε όλους τους τομείς, ε, γιατροί αλλά και απλοί άνθρωποι, έχουν στηρίξει με τη δράση τους αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Η Σίλβια Κώστα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξετίμησα πολύ και την παρέμβαση του Πρόεδρου Μουσκάτ και του κ. Μπόρκ για τι δεσμεύσει που ανελήφθησαν για να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα τη μετανάστευση. Το λέω σε Ευρωπαία και σαν Ιταλίδα. Πιστεύω ότι περιμένουμε πολλά από τη δική σα Προεδρία. Εξετίμησα πολύ και την μεγάλη συμμετοχή που έδειξε για το θέμα ο Επίτροπος ο κ. Πρέπει όλοι να πιστούμε γι' αυτό και χρειάζεται κατεπηγόντως να καλυφθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κυβερνήσεις όπως η ελληνική κυβέρνηση, να το πούμε με ειλικρίνεια, δεν καταφέρνουν να παρέμβουν επί θέματων ανθρωπιστικής ανάγκης, κατεπίγουσας ανάγκης που είναι εξαιρετική στη φύση της. Θα πρέπει λοιπόν, θα μεταφερθούν οι πρόσφυγες στα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και πιο πέρα όσον αφορά την έκκληση προς τις χώρες εκείνες που δεν ανταποκρίνονται στο καθήκον να υποδεχθούν τα ποσοστά των προσφύγων που του ανήκουν. Εμεί ζητήσαμε κυρώσει να επιβληθούν σε αυτέ τι χώρε ή να επιβάλλουμε κυρώσει μόνο για όταν παραβιάζονται οικονομικοί κανόνε. Θα πρέπει να ζητήσουμε να να θέσουμε και στην ε, συνείδησή μας το εξής ερώτημα. Ε, το λέω με ειλικρίνεια. Εχθέ η ακτοφυλακή Ιταλική είπε ότι η διάσωση των ζώων είναι όχι μόνο ηθικό αλλά και νομικό καθήκον. Αλλά το να σώζουμε τη ζωή επί της γης και στα όρια της ε, στερεάς γης έχει διαφορετική αξία. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσει διαφορετικά μηνύματα πάνω σε αυτό η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αν μιλούσα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, θα σας έλεγα τα χρήματα τα οποία θέλετε να δώσετε, δώστε τα μόνο στη Σερβία. Εκεί παγώνει οι άνθρωποι στο δρόμο και παγώνει και η καρδιά μας και εκεί θα πιάσουν τόπο τα χρήματα. Δεν παγώνουν στην Ελλάδα επειδή δεν έχουν διατεθεί χρήματα, έχουν διατεθεί και πολλά. Παγώνει, ε, παγώνουν οι άνθρωποι στα νησιά εξαιτία τη απίστευτη διοικητική ανεπάρκεια, τη κατασπατάληση πόρων μεταξύ ΜΚΟ και κυβερνήσεων και κυρίω παγώνουν εξαιτία σα, εξαιτία μα και εξαιτία των Ευρωπαίων πολιτικών. Η συσσόρευση στα νησιά γίνεται επειδή δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία με την Τουρκία από τη μεριά μας επειδή από το μάρτιο άνθρωποι περιμένουν την εξέταση της αίτησης ασύλου ώστε αυτοί που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες να μετακινηθούν στην εδωχώρα και να πάρουν άσυλο και άλλοι να επιστρέψουν στην τουρκία και χώρες που εξέτασαν ένα εκατομμύριο αιτήσει προσφύγων μέσα σε ένα χρόνο δεν μας δίνουν τους ανθρώπους που έχουν υποσχεθεί 800 ανθρώπους ειδικούς που έχουν υποσχεθεί όμως για να εξετάσουμε 15.000 αιτήσει. Αυτό ζητάμε από την Ευρώπη. Δεν ζητάμε ένα άλοθη, δεν ζητάμε χρήματα. Ζητάμε τους ανθρώπους μας που σχεθήκατε και αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Κύρκο. Ο κύριος Λόπεθ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα χιλιάδες πρόσφυγες ε, ε, υποφέρουν από το φρικτό κύμα κρύου στη Βαλκάνια και στην Ελλάδα με συνέπειες καταστροφικές και μάλιστα αυτό το υποφέρουν λόγω της δικής μας αδράνειας από ορισμένες κυβερνήσεις και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ε, παγωνιά χωρίς κατάλημα χωρίς ε, στέγη, χωρίς τρόφιμα. Ένα κύμα ψύχους που έχει ήδη προκαλέσει θανάτους, θανάτους ολόκληρη την Ευρώπη. Ανθρώπους που φεύγουν από τις χώρες τους γιατί ε, ε, ε έβρεχε βόμβες πάνω στα σπίτια τους. Κανένας δεν ξεκινά ένα τόσο επικίνδυνο δρόμο. Πρέπει να θυμίσουμε ότι 5.000 κόσμος πνίγηκε στη Μεσαίωγειο τον περασμένο χρόνο. Ε, κανένας δεν ξεκινά μια τέτοια πορεία αν δεν βρίσκεται σε πλήρη απελπισία. Ε, και ελπίζει να φτάσει σε μια ήπειρο που θα γίνει δεκτός. Σε αυτή η αδράνεια, η εν πάση περιπτώσει ανεπαρκή ε, ενέργεια θα έπρεπε να βαραίνει στι συνηθίσει μα. Γιατί πού είναι η ψυχή τη Ευρώπη ε, απέναντι στα όσα συμβαίνουν. Δεν μπορούμε πλέον να το ανεχθούμε λόγω τη αξιοπρέπεια και τη της δικαιοσύνη. Πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί με την συνεργασία τη εθνική κυβέρνηση ώστε να περάσουμε αυτό το κύμα ψύχους, να αποφύγουμε και άλλους θανάτους και κυρίως ε, να αποκαλύψουμε αυτούς που ήλπιζαν μόνο να βρουν ένα χώρο υποδοχής. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία ε, Μπιλμπάου Παραντίκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε οφείλουμε να εφαρμόσουμε τα επίγοντα μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα ψύχους, αλλά ε, κυρίως χρειαζόμαστε μια γενική απάντηση, μια σφαιρική απάντηση για να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση και να ανταποκριθούμε στις αξίες μας, αλλά να δημιουργήσουμε διαδικασίες που θα είναι ασφαλείς ε, ώστε να μπορούν να ζητήσουν ένα μήμα άσυλο αυτοί που το επιθυμούν. Η αλληλεγγύη των πολιτών έχει σαφώς εκφραστεί από πρωτοβουλία πρωτοβουλίε ανθρώπων ε, και οργανώσεων των πολιτών ε, αλλά και τοπικών οργανώσεων στο επίπεδο υποδοχής. Πρέπει λοιπόν να συνδεθούμε με αυτήν την ε, πολιτική και τη βούληση και να πιέσουμε τα κράτη που διστάζουν να υιοθετήσουν τέτοιου είδους δράσεις. Ε, το πρώτο του ταξίδι στο ε, εξωτερικό ε, του δικού μας Προέδρου ήταν να μπορέσει να γνωρίσει τους διαδρόμους πρόσβασης των προσφύγων και ελπίζουμε ότι θα μεταφέρει αυτές τις πολιτικές στην Ισπανία. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα έπρεπε να τρεπόμαστε ε, για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ε, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πόσο πολύ αποσύνδεση ε, αποσυνδέεται ο κόσμος από την Ευρώπη με, τα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και εσείς το γνωρίζετε το ξέραμε ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, όταν κανείς έχει τόσες χιλιάδες κόσμος, αυτό το λίμπο όπως είπε κάποιος, ε, ε, αυτό χειρότερο που μπορούσε να συμβεί συνέβη. Και συνέβη γιατί εμείς αυτό που μας απασχολεί στην Ευρώπη είναι να τους γυρίσουμε πίσω στην Τουρκία, να μην έρθουν εδώ. Όχι πώς θα του υποδεχτούμε, και αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα κράτη-μέλη που δεσμεύθηκαν με τι ποσοστώσεις για με την κατάσταση δεν τηρούν τι υποσχέσει του. και ειδικά η Ισπανία που ούτε στο 10% δεν έχει φτάσει, το 6% είναι. Είναι πραγματικά ντροπή αυτό που συμβαίνει και την ευθύνη φέρουν τα κράτη-μέλη. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι προ την Προεδρία τη Μάλτα, ειλικρινά. Τον άρχιστε σήμερα να μα λέτε για την εφαρμογή τη συμφωνία ε, με την Τουρκία, με τα όσα συμβαίνουν, ε, ε, νομίζω ότι είναι εκτό τόπου και χρόνου. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, και τώρα το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής ο κύριος ε, Επίτροπος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. για τη συζήτηση. Ήταν δύσκολη συζήτηση βεβαίως, γιατί όλοι εμείς αισθανόμαστε δυσάρεστα με την κατάσταση αυτή που επικρατεί και κανένας δεν είναι περήφανος. Ιδιαίτερα εξαιτία των ηθικών μας αξιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα θέλαμε να προσφέρουμε αξιοπρεπή διαβίωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε δεσμευμένοι στην στήριξη των εθνικών αρχών στις χώρες ιδιαίτερα που έχουν υπομειστεί το μεγαλύτερο βάρος. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ήταν σήμερα στη Λέσβο, ήταν σήμερα στην Ελλάδα, σε επαφή με τις τοπικές αρχές. Εγώ θα πάω το Σάββατο στην Σερβία και θα έχω επαχές, επαφές, θα συζητήσω με τις σερβικές αρχές, ιδιαίτερα για συνόδευτους ανήλικους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στο Βελιγράδι και με τα διάφορα μέσα που διαθέτουμε για την χρηματοδοτική στήριξη θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε κάποιες αδυναμίες. Το Σάββατο λοιπόν στη Σερβία θα ανακοινώσω επιπλέον χρηματοδότηση ιδιαίτερα για να στηρίξουμε τους εταίρους μας που εργάζονται για την αντιμετώπιση της ανθρωπικής κρίσης επιτόπου. Κανείς δεν πρέπει να συνεχίσει να παραμένει στο κρύο με αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες. Και συμφωνώ ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική και προκλητική περίοδο για την ευρωπαϊκή ιστηρία στέλνουμε μηνύματα προς τους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να παρέχουν πραγματικά στήριξη και βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν πράξεις και όχι λόγια. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες λοιπόν πιστεύω ότι θα κριθούμε θα κριθεί η δράση μας στο κατά πόσο είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους σας για τη στήριξή σας, γιατί σήμερα είδα ότι είστε διατεθειμένοι να μας στηρίξετε για να συνεχίσουμε σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο. Και βεβαίως άσχετα με το πόσο επίγουσα είναι αυτή η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την επίγουσα κατάσταση, οι προκλήσεις είναι πολλές, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση με μακροπρόθεσμο τρόπο αυτών των καταστάσεων. Η Προεδρία της Μάλτας θα πρέπει να συνεχίσει αυξάνοντας τον αριθμό των ανθρώπων που θα μπορούν να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και από την Ελλάδα. Χρειάζονται ειδικοί για θέματα ασύλου, οι οποίοι να στηρίξουν τις αρχές των χωρών αυτών. Και εδώ συμφωνώ πολύ με τον κύριο Κύρκο. Το θέμα λοιπόν των ειδικών για θέματα ασύλου, οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται επιτόπου και να στηρίζουν τις εθνικές αρχές των χωρών αυτών, δεν έχει καλυφθεί. Μόνο η μισή από αυτούς που έχουν ε, ζητηθεί από τις χώρες, ε, την Ελλάδα και την Ιταλία, έχουν φτάσει. Παραδέχομαι λοιπόν εδώ ότι βεβαίως υπάρχουν και κάποια επίμαχα σημεία στην συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Την ίδια ώρα όμως, μέσω αυτής της συμφωνίας μπορέσαμε να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό αυτών που έφταναν στην Ευρώπη. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω κάτι. Αυτή η προσφυγική κρίση δεν είναι εθνικό θέμα της Σερβίας, της Ιταλίας ή της Ελλάδας ή της Ισπανίας. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η λύση δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική ευρωπαϊκή. Γι' αυτό και επιμένουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση. Γι' αυτό και ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα να μας ε, βοηθήσει. Πρόκειται την ίδια ώρα για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Πρόκειται για μια παγκόσμια ευθύνη. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάποια άλλα σημεία, σύμφωνα απολύτως με τη Λίντα, Α, για το θέμα των vouchers για τα τρόφιμα. Τα κουπόνια είναι κάτι το καθοριστικό για την αξιοπρέπεια των προσφύγων. Είναι μία από τις τέσσερις σημαντικότερες προτεραιότητες μου στην Ελλάδα. Και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και για μας αυτό θα πρέπει να είναι η βάση αυτής της δράσης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στους καταβλισμούς προσφύγων. Η εμπειρία μου, αλλά και οι αξιολογήσεις που προέρχονται από τους συνεργάτες μου, μου δείχνουν ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο οικονομικό να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο τροφοδοσίας σε σχέση με άλλα συστήματα όπως αυτό παραδείγματο χάρη που χρησιμοποιείται σήμερα για την τροφοδοσία στην Ελλάδα. Επίσης, στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο και την τοπική οικονομία, την τοπική αγορά. Γι' αυτό και στην Τουρκία χρησιμοποιήσαμε το σύστημα ESSN για ένα εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες που διαμένουν στην ε, Τουρκία. Ο Υπουργός ε, Μεταναστευτικής Πολιτικής ε, της Ελλάδας, ο κ. Μουσάλας, ανακοίνωσε και επίσημα την επιλογή αυτού του νέου συστήματος τροφοδοσίας των προσφύγων μέσω των κουπονιών και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει και πρέπει να γίνει με μεγάλη ταχύτητα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράες, πρόεδρε Μωράες, για τα πολύ θετικά σας λόγια. Ναι, υπάρχει χρηματοδοτική δυνατότητα και εμείς θα στηρίξουμε τη δημιουργία νέων καταβλισμών, νέων δυνατοτήτων στέγασης και φιλοξενίας προσφύγων Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος προσπαθούν να βρουν λύσεις. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν ε, σε καθημερινή βάση λύσεις ε, για τη φιλοξενία των προσφύγων, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να το βελτιώσουμε το σύστημα φιλοξενίας προσφύγων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάτι που πολλοί από εσάς ε, είπατε. Μιλήσατε για την μεταφορά των μεταναστών και των προσφύγων από τα νησιά της ε, Ελλάδας στην ενδοχώρα. Και βεβαίως μετά από πολλές ε, συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές πήραμε την απόφαση να μεταφέρουμε τουλάχιστον τις ευάλωτες ομάδες ε, ανθρώπων έτσι ώστε να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης διαβίωσής τους. Και είδαμε στην ενδοχώρα, στην υπηρετική Ελλάδα, ότι υπήρχαν δυνατότητες αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Πολλοί πρόσφυγες, οι οποίοι βρέθηκαν σε καταβλισμούς ε, με ικανοποιητικές συνθήκες, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης ή ε, της Αθήνας. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα τροφοδοσίας μέσω των ε, κουπονιών μέχρι τον Μάρτιο στην Ελλάδα, εάν καταφέρουμε να μεταφέρουμε περισσότερους πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου στην υπηρετική Ελλάδα, νομίζω ότι η κατάσταση σαφώς και βελτιώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για τη στήριξή σας, για τη βοήθειά σας, για αυτό το πάρα πολύ δύσκολο θέμα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ομιλία σας αυτή εκ μέρους του Συμβουλίου. Ο κ. Μπόρκ, ο κ. υπουργό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για αυτά που είπαν, για τις απόψεις τους. Ως Προεδρία πρέπει να πω ότι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται. Γνωρίζουμε τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Ελλάδα και στη Σερβία. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ανέφερε ποια μέτρα λαμβάνονται, ποιοι πόροι είναι στη διάθεσή μας, τι μέσα διαθέτουμε. Ως Προεδρία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις προς όφελος της αξιοπρέπειας των μεταναστών και των προσφύγων. Στο κάτω-κάτω δεν ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο έτσι από καπρίτσιο. Ήρθαν εδώ διότι προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους, από διώξεις στις πατρίδες τους. Όμως, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω κάτι. Η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες που αναφέρθηκαν, από τους αξιότιμους ευρωβουλευτές έχουμε αυτή την εμπειρία, διότι τα τελευταία χρόνια όχι μόνο τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα χρόνια το ζήσαμε αυτό. Μόνοι μας, ίσως να μην είχαμε ξανακούσει τις συζητήσεις αυτές που έγιναν εδώ στα θεσμικά όργανα, αλλά από μόνοι μας, από πρώτο χέρι, ξέραμε ποια είναι η κατάσταση. Κάθε μέρα πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς την κατάσταση κατά την οποία πρέπει να σώσει ανθρώπους στη θάλασσα, Επίσης, πρέπει να υποδεχθεί αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να τους εντάξει στην κοινωνία της κάθε χώρας. Ο Πρωθυπουργό μας μας το είπε σαφώς σήμερα το πρωί. Πρέπει να εργαστούμε περισσότερο στο Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όσα συμφωνήθηκαν εφαρμόζονται. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στη μετεγκατάσταση. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να δούμε πώς εκείνες οι χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με την ποσόστοση που δεσμεύτηκαν να πάρουν, πώς αυτές οι χώρες μπορούν να κάνουν περισσότερα. Όμως θα πρέπει επίσης να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα σύνορά μας. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτά που συμφωνήσαμε όταν προσφέραμε μια βάση, μια πλατφόρμα για, διοργανώσαμε την ε, Σύνοδο κορυφή της Βαλέτα πάνω από, εδώ και πάνω από ένα χρόνο και τότε όσον αφορά την εξωτερική πτυχή συναντήσαμε όχι μόνο τους Ευρωπαίους συναδέλφους αλλά και τους Αφρικανούς συναδέλφους. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε συνάντηση υψηλού επίπεδου για να συζητήσουμε την επιτευχθήσα πρόοδο από όλες τις πλευρές και πώς οι επενδύσεις, τα χρήματα που δώσαμε ε, χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να αλλάξει η παράνομη δραστηριότητα στην Αφρικανική Ήπειρο. Να γίνουν όλα πιο θετικά. Θα εργαστούμε σκληρά, παρόλο που γνωρίζουμε ότι σε έξι μήνες δεν μπορούμε να βρούμε και όλες τις λύσεις, όμως θα συνεχίσουμε να προοδεύουμε για να δείξουμε ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε εξίσου τις ευθύνες. Ξανά λέγω ότι ξέρω τι είναι να αντιμετωπίζει κανείς μόνος του τα προβλήματα. Γι' αυτό ως Προεδρία θα καταβάλουμε προσπάθειες, θα συνεχίσουμε το διάλογο με τις χώρες για να πετύχουμε πρόοδο για καλύτερο επιμερισμό των ευθυνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πρώτη αυτή ευκαιρία που είχα να μοιραστώ τις απόψεις μου μαζί σας και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε παρομοίως τη συνεργασία μας και στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που μιλήσατε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτά που μας είπατε κύριε Υπουργέ, για τη δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημαντικό θέμα.